We'll just hold it present for a moment. Yeah. Připomínka k jednání, prosím. Τι θέλατε διαδικαστικό, έχετε το λόγο. Το μικρόφωνο σας δεν ήξερα. Ήδη συζητήθηκε Και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξή. Γνωρίζετε ότι στην Ολομέλεια τέθη αυτό το θέμα από τον κύριο Σαλαφράγκα. Εμείς το συζητήσαμε με την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και με βάση το άρθρο 140 παράγραφος 2 προκύπτει το εξής. Η πρόταση για το κατά πόσον θα συζητηθεί το θέμα ε, θα γίνει με ονομαστική κλίση. Μπορείτε λοιπόν να τοποθετηθείτε ακριβώς λόγω της ονομαστικής κλίσης και εάν υπερψηφιστεί η πρόταση θα συνεχιστεί η συζήτηση. Αλλιώς το θέμα αυτό ε, θα περάσει χωρίς συζήτηση. Επαναλαμβάνω, ξαναψηφίζουμε με ονομαστική κλίση επί του θέματος. Διακόπτω όμως τώρα μισό λεπτό ε, για διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, Θέλω πολύ σύντομα να πω το εξή. Βεβαίω είναι κάπω περίεργο το να ερχόμαστε εδώ σε μία συζήτηση, περιμέναμε να γίνει συζήτηση και τελικά τι γίνεται, καταργείται αυτή η συζήτηση. Αυτό είναι το ένα περίεργο. Το δεύτερο είναι ότι προφανώ ε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε σωστά όπω το προτείνονται εσεί κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο οι συνάδελφοι έχουν μαζί του την κάρτα του. Αν ε, ψηφίσουμε να, ε, θα έπρεπε να υποθεί ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία και όχι τώρα που έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση να μας λέτε ξαφνικά ότι θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Γιατί αν ψηφίσουμε, εγώ παρακαλώ να ψηφίσουμε με ανύψωση ε, των ε, χεριών και όχι ηλεκτρονικά. Αυτό επιθυμώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, να σας πω το εξής, ότι Εχθές το είχαμε πει στις πολιτικές ομάδες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρα μπορούσατε να προετοιμαστείτε. Πριν λοιπόν ψηφίσουμε υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση γιατί δεν θέλω να αποκομίσετε την εντύπωση ότι εγώ θέλω να επηρεάσω καθιονδήποτε τρόπο τη συζήτηση. Όλα που γίνονται τώρα τα έχουμε συζητήσει με την νομική μας υπηρεσία. Εγώ θα ήθελα απλώς να μας διευκρινίσετε το πώς θα ψηφίσουμε. Και τι, θα ψηφίσουμε. Ψηφίσουμε και όταν θα κάνουμε τη ζήτηση ή όχι. Για να ξέρουμε. Πώς θα ψηφίσουμε. Επομένω, το ξαναλέω. Θα ψηφίσουμε αφού όλοι τοποθετήθηκαν. Okay. Επαναλαμβάνω, λέει ο Πρόεδρος, θα σας εξηγήσω πώς έχουν τα πράγματα. Και συγχωρήστε με. Αυτοί που θα ψηφίσουν υπέρ σημαίνει ότι επιθυμούν να διακόπτει. Διακόπτει prosím vás jedná se o natolik vážné hlasování že je třeba trošku mírnit emoce. ještě Είναι πάρα πολύ σημαντική η ψηφορία αυτή, λέει ο Πρόεδρο. Ε, ξέρω, ε, γι' αυτό το λόγο και ε, έχουν ανάψει τα πνεύματα. Θα ψηφίσουμε σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του κανονισμού μας. Υπάρχει η πρόταση. Το πρώτο σημείο της συζήτησης όσον αφορά την παραγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου, δηλαδή πρόκειται για το σημείο το οποίο αφορεί το Γουαντάναμο και του απεργού πείνα, αυτό να ε, εγκριθεί χωρί συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αυτό το αίτημα. Είναι σαφέ. Ωραία. Οπότε τώρα ψηφίζουμε. Με ψήφισαν όλοι. Πέρασε ο the members voting? Members voting 44. In favour 25. Against 19. Yeah. So it's carried. It was carried. Εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς δεν θα γίνει συζήτηση. We now come to the... Yeah. Yeah. So this one